Μία ανακοίνωση να σας κάνω. Ο κύριος Κάλλος Χιμένες Φιλαρέχο μου ανακοίνωσε την ε, παρέτησή του ε, από την 1η Αυγούστου του 2014. Και έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο ανακοινώνει ότι όσον αφορά την ε, θέση αυτή του κυρίου Κάλλος Χιμένες Μιναρέχο η θέση αυτή χειρεύει και θα ενημερώσει σχετικά το κράτος μέλλον. Και όσοι ταξιδεύετε σας εύχομαι καλό ταξίδι, καλές διακοπές, εύχομαι όμως να φύγετε και όσο το πιο γρήγορο γίνεται έτσι ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας που είναι επεξηγήσεις σε ψήφου. Περνάμε λοιπόν στις επεξηγήσεις ψήφου. Παρακαλώ συνάδελφε διαδικαστικό, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω πλήρη κατανόηση για το γεγονό ε, προηγουμένω. Δεν θέλατε να συνεχίσετε αυτά που ελέγχθησαν. Μόνο που ήθελα να πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με τον τρόπο που διευθύνετε τη συζήτηση. Τα κάνετε πάρα πολύ καλά και θα προέτεινα σε όλου του συναδέλφου να είναι λιγάκι πιο συγκεντρωμένοι και αν το κάνουν αυτό, τότε νομίζω ότι θα εργαζόμαστε θαυμάσια. Πρόεδρος, περνάμε τώρα λοιπόν στις επεξηγήσεις ψήφων, καταρχήν όσον αφορά τις τροπολογίες για την κατάσταση στην Ουκρανία. Και ξεκινάει ο συνάδελφο κύριος Τάνοκ που μιλάει εξ ονόματος της πολιτικής ομάδας και για το λόγο έχει δύο λεπτά στη διάθεσή του. Η ομάδα μας θεωρεί ότι η αποτελεσματική νίκη του Πρόεδρου Ποροσέγκο, ο οποίος